Περνάμε στις επεξηγήσεις ψήφου. Έχουμε πολλές αιτήσει. Δεν μπορούμε όμως να καθυστερήσουμε πέρα από τις 14 και 45 γιατί οι υπηρεσίες πρέπει να έχουν χρόνο να προετοιμάσουν την αίθουσα πριν από την έναρξη της επόμενης συνεδρίασης στις 3. Όσοι δεν μπορέσουν να πάρουν το λόγο σήμερα, αύριο μετά τις ψηφοφορίες θα έχουν αυτή την ευκαιρία. Περνάμε λοιπόν στην έκθεση Νικολάη. Ο κύριος Ανάν έχει το λόγο. Κύριε Αντιπρόεδρε, ένα πράγμα έχω να πω. Ε, μετά από χρόνια που βλέπω την υποκρισία και τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά, δεν